Κυρίε Κυρίες και κύριοι, θα συνεχίσω στα Ουγγρικά που είναι και η μητρική μου γλώσσα και ελπίζω να είναι πολλοί που μιλούν την Ουγγρική και να με καταλαβαίνουν, αλλιώς έχουμε και υπηρεσίες διερμηνίας, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να απευθύνω θερμό χαιρετισμό προς τον Πρόεδρο, που, μου, που με επέπληξε γιατί στην αρχική μου ομιλία υπερεύει το χρόνο αγόρευσης και με μάλωσε ο πρόεδρος. Είχα 7 λεπτά ως πρόεδρος που παρουσίαζε το πάνελ ε, και εγώ έκανα κάποια κατάχρηση χρόνου. Οπότε πάμε κατευθείαν στη στρογγυλή τράπεζα. Θα δώσουμε το λόγο στην πρόεδρο ε, της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, Έχουμε επιφανείς καλεσμένους που θα μας μιλήσουν για το θέμα της Τρογγυλής Τράπεζας. Θα μιλήσουμε για την ανάπτυξη, την απασχόληση. Έχουμε πολλούς καλεσμένους που θα αγγίψουν στις διαφορετικές πτυχές του θέματός μας που είναι η προσέλκυση των επενδύσεων και η βελτίωση του επιχειρηματικού κλιμάτος. Και επίσης έχουμε μαζί μας μια πολύ συμπαθητική και εξαιρετικά δραστήρια επίτροπο, πολύ οικία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την κυρία Τάισεν, που θα λάβει και αυτή μέρος στη Στρογγυλή Τράπεζα εκ μέρους Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Mm. Έχετε το λόγο λοιπόν πρώτα εσείς κύριε Επίτροπε. Αγαπητέ Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, εξοχότητες κυρίες και κύριοι, είμαι πασιχαρής ε, για τη συμμετοχή μου εδώ σήμερα ε, για να συζητήσουμε πώς θα προσελκύσουμε επενδύσεις και θα βελτιώσουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον σε ένα από τους στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας. Ο τουρισμός και οι συναφείς δραστηριότητες απασχολούν 12 εκατομμύρια πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή το 22% των θέσεων απασχόλησης στον τομέα των υπηρεσιών και μάλιστα ε, ε, δημιουργεί 5 ε, εκατομμύρια, μάλλον θα δημιουργήσει κατά πάσα πιθανότητα 5 εκατομμύρια νέε θέσει απασχόληση την επόμενη δεκαετία με βάση κάποιες προβλέψεις. Οπότε ο κλάδος αυτός προσφέρει προτεραιότητες σε ανθρώπους κάθε ηλικία και, δεξιότη, και δεξιότητες. Και μάλιστα 20% είναι μέχρι 24 χρονών, 58% είναι γυναίκες και περίπου 50% είναι ε, μετανάστες ε, εργαζόμενοι. Οπότε είναι σημαντικός, σημαντική πύλη εισόδου ε, στην αγορά εργασίας και κινητήριος μοχλούς ανάπτυξης. Επίσης, εξαρτάται από τους εργαζόμενους ο τουρισμός, ειδικευμένου κυρίως, και οι δεξιότητες αυτές αποκτούνται με εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση, που μερικές φορές όμως δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου. Επίσης, ε, ο τουριστικός κλάδος έχει και ένα πρόβλημα εικόνας, ε, γιατί οι τουριστικές δραστηριότητες ε, θεωρούνται πολλές φορές εποχιακές και χωρίς προοπτική σταδιοδρομία ή χαμηλή αμοιβή. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερη συνεργασία μεταξύ του κλάδου του τουρισμού, των δημοσίων αρχών και κρατικών φορέων και των πανεπιστημίων ή των φορέων παροχή εκπαίδευση, ώστε να προσαρμόσουμε το σχολικό πρόγραμμα στις πραγματικές ανάγκες αγοράς για να, μην, για να γίνει πιο ελκυστικός, πιο βιώσιμος και πιο ανταγωνιστικός ο τουρισμός. Ο τουρισμός μάλλον, μάλιστα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι από τους ε, πιλωτικούς κλάδους ε, της στρατηγικής για την ε, διακλαδική συνεργασία και περιλαμβάνεται και στο θεματολόγιο μας για τις δεξιότητες. Και μάλιστα έχουμε ένα, μια σύμπραξη της Κοφιντούστρια με εταίρους από το τουριστικό κλάδο 10 χωρών μελών. Και μάλιστα ε, χορηγούμε περίπου ε, επιδοτήσεις 4 εκατομμυρίων ε, ευρώ προκειμένου να λυθούν βασικές ανάγκες δεξιοτήτων και να χαράξουμε μια στρατηγική ευρωπαϊκών δεξιοτήτων για τον τουρισμό, να αναβαθμίσουμε, να αναπτύξουμε τα σχολικά προγράμματα και να προωθήσουμε την ελκυστικότητα του κλάδου ε, και επίσης να προσφέρουμε δυνατότητα ε, απόκτησης επαγγελματικής πείρας ε, και σε φοιτητές και σε ανέργους. Αυτό θα δώσει μια όθηση στον τουρισμό, γι' αυτό σας παροτρύνω να λάβετε και εσείς μέρος για να διαμορφώσουμε αυτή τη στρατηγική μας για τον τουρισμό. Επίσης, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σε μια νέα πρωτοβουλία, το έρασμο για τους επαγγελματίες, που τον επόμενο, τον επόμενο βήνα θα εγκαινιάσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για μια νέα εκδοχή του γνωστού προγράμματος Έρασμος και μάλιστα το Έρασμος για τους επαγγελματίες ε, θα είναι προσιτό σε νέους από διάφορα υπόβαθρα 400 εκατομμύρια ευρώ είναι ο προπολογισμό ε, για το 2018 με 2050. Θα δώσουμε 50, την ευκαιρία σε 50.000 ε, ασκούμενους και φοιτητές να ε, παρακολουθήσουν ε, περίοδους άσκησης και στην αλλοδαπή. Οπότε αυτή η διασυνοριακή ευκαιρία που τους δίνουμε πιστεύουμε ότι θα τους δελεάσει και έτσι θα έχουμε και εταιρικέ σχέσεις τουρισμού με ενδιαφερομένους που είναι παρόντες σήμερα αλλά και με ε, φορείς παροχής κατάρτισης και εκπαίδευση. προκειμένου να αξιοποιηθεί στο έπακρο αυτή η νέα πρωτοβουλία, το Έρασμος για τους επαγγελματίες, Έρασμος προ- Επίσης, έχουμε νέα δημοσιονομικά κονδύλια για τις, για τις ασκήσεις και σε συνεργασμό με το τομέα παραγωγής τροφίμων, γεωργίας και τουρισμού και στα πλαίσια του γενικότερου ε, της γενικής οργάνωσης που κατηλείπτει τους ε, εστιατόρες, ξενοδόχους κλπ. Επίσης, σας ευχαριστώ θερμά για την υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας ε, για τις ασκήσεις, γιατί πραγματικά ε, ποιοτικέ ε, περίοδοι άσκησης ε, θα αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο για ποιοτικέ θέσει απασχόληση. Και είμαι πεπισμένη ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να μην φυσιστούμε προσπαθειών προκειμένου να προωθήσουμε και να στηρίξουμε τέτοιε ποιοτικέ θέσει άσκηση. Και ελπίζω να συμβάλλετε με την ΕΦΤΑ και τη ΧΟΤΡΕΚ σε αυτή την αναβάθμιση των θέσεων άσκηση. Επίσης, τον Νοέμβριο θα οργανώσουμε τη δεύτερη ετήσια εβδομάδα για την εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, ΒΕΤ, με εκατοντάδες εκδηλώσεις και σεμινάρια σε όλη την Ευρώπη. Και ελπίζω να έχουμε πολλές εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες και του τουριστικού κλάδου και ελπίζω να συμβουλευτείτε το, την ιστοσελίδα ή την, το επιτελείο ΒΕΤ και τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης που είναι αρμόδια για τα θέματα αυτά προκειμένου να ενημερωθείτε για το πώς θα ε, προωθήσετε και εσείς τις δικές σας δραστηριότητες και πώς θα εμπλακείτε στο, στην πρωτοβουλία αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε δεξιότητες ώστε να αποκτήσει ο τουρισμός πραγματικά πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση αυτής της εβδομάδας για την επαγγελματική κατάρτιση και παιδεία. Σας ευχαριστώ, σας εύχομαι καλή τύχη, ευχαριστώ για την προσοχή Λυπούμε λόγω της καθυστέρησης, ε, έχω ανηλυμένη υποχρέωση, οπότε δεν θα μπορέσω να παρακολουθήσω την συνέχεια των συζητήσεων, αλλά σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε κυρία Επίτροπε, κυρία Τέισεν. Ήταν παρόλα αυτά πολύ χρήσιμη παρουσίαση εδώ. Μα ε, μας παρουσιάσατε τις σκέψεις για τον τουρισμό και μας ζητήσατε την αρρωγή μας προκειμένου να στηρίξουμε τον κλάδο. Σας ευχαριστώ. Ξέρω ότι Πολύ γεμάτο το πρόγραμμά σας. Καλή συνέχεια. Επόμενος ομιλητή είναι ο κύριο Βάσιλ Χούντακ, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ελπίζω να μας φέρει χαρμόσυνα νέα για τον τουρισμό. Κύριε Χούντακ, έχετε το λόγο. you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για, την, για τα καλά σας λόγια ε, κυρία Επίτροπε, κύριε Υπουργέ, ξεχότατα μέλη του Κοινοβουλίου, φίλοι του τουρισμού, να σας πω ότι είναι χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να εορτάσουμε αυτή την ημέρα του τουρισμού και για να στηρίξουμε και την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών. Θεωρώ ότι είναι μοναδική ευκαιρία για μας ε, το να συζητήσουμε για το πόσο ο τουρισμός μπορεί να καταστεί ακόμα σημαντικότερος για την ε, ευρωπαϊκή οικονομία. Πράγματι, ακούσαμε πάρα πολλά για το πόσο σημαντικός είναι ο τουρισμός. Είναι το μα της Ευρώπη, Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας, του πολιτισμού μας και παράλληλα ε, ποτέ δεν τελειώνουν αυτά που μπορούμε να κάνουμε για να στηρίξουμε τον τουρισμό. Και εξάλλου κι όλοι μας είμαστε τουρίστες όλοι ταξιδεύουμε ε, με τις οικογένειές μας και όχι. Ε, έτσι λοιπόν σήμερα προσφέρεται η ευκαιρία πώς μπορούμε να κάνουμε περισσότερα για να στηρίξουμε αυτό το σημαντικό κλάδο της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όπως αναφέρθηκε ήδη, εγώ εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Είναι η τράπεζα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που ε, κυβερνάται από τα 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ο μεγαλύτερος ε, πολυμερής ε, χρηματοδοτικός οργανισμός της Ευρώπης. 84 δις ήταν επενδύσεις μας πέρσι. Τα τελευταία 50 χρόνια 30 εκατομμύρια πήγαν στον τουρισμό, 30 δις με συγχωρείτε, πολλά, αλλά δεν είναι αρκετά για μας, είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο τουρισμός είναι ένα σημαντικό κομμάτι της οικονομικής ανάπτυξης Ευρώπης ε, και πολύ συχνά δυστυχώς ε, υποτιμάται, αλλά ε, πρέπει να το πούμε, έτσι είναι. Ο τουρισμός είναι η τρίτη σημαντικότερη κοινωνική δραστηριότητα της Ευρώπης και βοηθάει ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ευημερία της. Η Ευρώπη είναι ο μεγαλύτερος τουριστικός προορισμός στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, όπως είπε και η κυρία Επίτροπος, ε, δημιουργεί θέσεις απασχόληση ε, προσφέρει νέες ευκαιρίες για τους νέους σε χώρες και διάφορες περιοχές της Ευρώπη. Η συνεισφορά του τουρισμού στην οικονομία είναι περίπου στο 10% του ΑΕΠ. Σημαντικό το ποσοστό αυτό και τα, οι αριθμοί είναι πολύ εντυπωσιακοί. Ο τουρισμός γίνεται όλο και περισσότερο πηγή καινοτομίες, δεύτερα ας πούμε εταιρείε, όπως, όπως, είναι η Airbnb που δυστυχώς δεν είναι ευρωπαϊκή αλλά από τον τουρισμό προέκυψε. Υπάρχει λοιπόν μια σημαντική πρόκληση. Πώς θα μπορέσουμε να συνδυάσουμε την ιστορία, τον πολιτισμό με τον νεοτερισμό, πώς μπορούμε να συνδυάσουμε την ε, πολυμορφία με ένα συγκριτικό πλεονέκτημα της Ευρώπης. Άρα είναι σημαντικό το πώς χρηματοδοτείται και ο τουρισμός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με διάφορους τρόπους. Ένας εξ αυτών είναι με άμεση χρηματοδότηση των ξενοδοχείων και με ενδιάμεσους. Ενδιάμεσους τώρα είναι οι τράπεζες, ε, διάφοροι οργανισμοί. Παραδείγματος χάρη έχουμε χρηματοδοτήσει ένα δάνειο ε, για την ε, αναβάθμιση των ξενοδοχείων στην Ισπανία. Επίσης έχουμε προσφέρει περίπου ένα δις ευρώ για την ανάπτυξη τουρισμού, κυρίως για την υποδομή και για πολιτιστικές υποδομές. Ε, πρόκειται για δάνεια σε πόλεις, ε, σε πολλούς τομείς. Έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τις ε, ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στην Ουγγαρία, περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ για το, την αναμόρφωση περιοχής στην Ισπανία. Στην κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη πολύ συχνά Είμαστε συγχρηματοδότης από κοινού με τα διευθυντικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν αυτούς τους οργανισμούς, αυτή τη μορφή χρηματοδότηση στην μεικτή και μετά το 2020 αυτός κατά πάσα πιθανότητα, αυτό το blending, θα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς τρόπους για το πώς χρηματοδοτούνται τα έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, χρηματοδοτούμε επενδύσεις σε διάφορα σημαντικά και ουσιαστικά μέρα της Ευρώπης ε, σε μουσεία μεταξύ άλλων. Στηρίζουμε λοιπόν τον τουρισμό, προσφέρουμε απευθείας δάνεια αλλά και δάνεια σε τράπεζες. Ένα μεγάλο κομμάτι των επενδύσεών μας γίνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τυχαίνει και αυτές να εμπλέκονται με τον τουρισμό. Από το 10 μέχρι το 16 6 δις ευρώ δόθησαν για να στηριχθούν ΜΜΕ, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στον τουρισμό. Αναφέρθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων διαχειρίζεται και το Ευρωπαϊκό Ταμείο για Στρατηγικές Επενδύσεις, ε, ένα κομμάτι του προγράμματος Juncker και είναι μια προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να, ε, να, να δώσει νέα όθηση στην οικονομική ανάκαμψη στην Ευρώπη. Ίσως να μην έχουμε κάνει αρκετά ένα καλό παράδειγμα ε, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΦΣΥ είναι η χρηματοδότηση τουριστικής εγκατάστασης Μπαλαμάρ στην Κροατία. Ε, αυτή η χώρα εξαρτάται πάρα πολύ από τον τουρισμό και θέλουμε να κάνουμε και άλλα, να χρηματοδοτήσουμε φορείς του ιδιωτικού τομέα, κυρίως σε ε, ε, περιοχές που εμπίπτουν σε στόχους ε, συνοχής και σύγκλησης. Γιατί δεν κάναμε περισσότερα, υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι, όπως το ότι ο τουρισμός είναι ένας ε, τομέας ε, με πολλές μεταπτώσεις ε, και μερικές φορές υπάρχουν και αντιδράσεις από κράτη-μέλη στο να χρηματοδοτηθούν ξενοδοχεία πέντε αστέρων. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά εμείς ως τράπεζα είμαστε στρατευμένοι έναντι του τουρισμού. Έχουμε μια νέα στρατηγική και όσοι ενδιαφέρονται τους καλώ ανεπιφύλακτα να έρθουν να συζητήσουμε για νέα προγράμματα. Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή μου, θέλω να υπογραμμίσω, δεν είμαστε μόνο ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός, προσφέρουμε και συμβουλές και με μεγάλη μας χαρά να συνεργαστούμε με κυβερνήσεις, με τοπικούς φορείς, αλλά και με ιδιώτες για να διαρθρώσουμε προγράμματα τα οποία ε, θα είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Να μας αντιμετωπίζετε ως εταίρος στην αποκαλούμενη επανάσταση του τουρισμού Είμαστε στη διάθεσή σας, θέλουμε να συνεργαστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ και για την προσοχή σας. Και εμείς ε, σας ευχαριστούμε. Θέλω να πιστεύω ότι οι πληροφορίες που δώσατε ήταν πολύ ενδιαφέρουσες ε, για τους προσκεκλημένους μας. Η επόμενη έρχεται από τη Βουλγαρία η ομιλήτριά μας είναι ε, ιδιαίτερα δραστήρια, πολύ δραστήρια υπουργό Τουρισμού, από τις πιο δραστήριες ε, στην Ευρώπη και αν θυμάμαι καλά, πριν από δύο εβδομάδες ήμασταν στο ίδιο πάνελ στην Κίνα, στην ε, Γενική Συνέλευση του ΠΟΑ. Γνωριζόμαστε λοιπόν πάρα πολύ καλά και ελπίζω ότι θα μπορέσει η κυρία Αγγέλκοβα να περάσει σημαντικά μήνυματα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, εξοχότητες, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνάδελφοι και φίλοι του Ευρωπαϊκού Τουρισμού. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που συμμετέχω σε αυτή την εκδήλωση υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με αντικείμενο την ε, Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Συγχαρητήρια σε όλους, σας εύχομαι καλή επιτυχία καλή συνέχεια ώστε ο τουρισμός μας να πάει ακόμα πιο καλά και να γίνει ακόμα πιο αηφόρος. Είναι στρατηγικό τομέα τη οικονομία μα ο τουρισμό στην Βουλγαρία αλλά και σε άλλε χώρε. Είναι πηγή ανάπτυξη και θέσεων απασχόληση. Το Παρίσι, η Ρώμη, η Βαρκελόνη, πάρα πολλέ πόλει στην Ευρώπη είναι μέσα στου πρώτου τουριστικού προορισμού του κόσμου. Χάρη στο φυσικό μα τοπίο, στι πολιτιστικέ και φυσικέ ομορφιέ, η Ευρώπη δέχεται επισκέψει εκατομμυρίων πολιτών, αλλά και η Βουλγαρία το ίδιο. 8 ε, εκατομμύρια 200 χιλιάδες τουρίστες δεχτήκαμε ε, πέρσι. Το πιο σημαντικό είναι ότι 3 δις 200 εκατομμύρια ευρώ ξοδεύτηκαν στη Βουλγαρία από τουρίστες και μέσα στον κλάδο του τουρισμού, αμέσως και εμέσως. Και γι' αυτό η κυβέρνησή μας θεωρεί ότι ο τουρισμός είναι στρατηγικό, ε, είναι στοιχείο κλειδί της οικονομίας μας. Έχουμε υιοθετήσει στρατηγική, οδικό χάρτη και σχέδιο δράσης για τον τουρισμό. Ε, θέλουμε ο τουρισμός οριζόντια να ενταχθεί ε, σε όλες τις δράσεις όλων των Υπουργείων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες, την ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων, μια βασική αξία για τις Ευρωπαϊκές Ένωσης. Όμως η συνδεσιμότητα και οι υποδομές είναι κάτι πολύ σημαντικό για την οηφόρο ανάπτυξη του τουριστικού τομέα. Η κυβέρνηση της Βουλγαρίας αξιοποιεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια για να εξυγχρονίσει το οδικό δίκτυο, το δίκτυο των υποδομών και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις υποδομές μας και τις συνδέσεις μας με, τους, με τις γειτονικές χώρες, Ελλάδα ε, μεταξύ άλλων. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικό σημαντικά για να έχουμε καλύτερη ανάπτυξη. Οι υποδομές οι αεροπορικές είναι εξίσου σημαντικές και η συνδεσιμότητα αυτών και θέλουμε να προωθήσουμε τα ΣΔΙΤ. Και προωθούμε επίσης τις, τους διάβλους μεταφορών και επικοινωνιών μέσα από το Δούναβι αλλά και μέσα από τον Πόντο. Είναι μια χώρα που ε, ε, η Βουλγαρία που είναι μέλος στην ομάδα τη συντονιστική για τις χώρες του Ευξήνου Πόντου και η ομάδα εργασίας θα ασχοληθεί στην επόμενη συνεδρίαση ε, με το θέμα της ανάπτυξης και της προώθησης της τουριστικής δραστηριότητας στη Μαύρη Θάλασσα. Στη Βουλγαρία τα τελευταία χρόνια οι τουρίστες από το εξωτερικό έρχονται με πολύ και είναι περισσότεροι από τις δυνατότητες καταλήμματων. 6,2 εκατομμύρια τουρίστες δεχτήκαμε από το εξωτερικό, αύξηση 8% μέσα σε ένα χρόνο. Επομένως, το Υπουργείο Τουρισμού θέλει να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις για ε, ξενοδοχεία. Για ξενοδοχεία. Και Θέλουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις στις ξενοδοχειακές υποδομές, όχι μόνο στα θερινά και στα χειμερινά, ε, στα θερινά, και στα χειμερινά θέρετρα, αλλά και στα σημεία και στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς, σε αυτές τις τοποθεσίες και τις πόλες. Πρέπει να συνεργαστούμε πιο στενά, και να πάμε προς την αηφόρο ανάπτυξη. Και γι' αυτό βασική προτεραιότητα είναι να μειώσουμε το διοικητικό φορτίο και για τους πολίτες και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουμε μια μονοαπευθυντική θηρίδα για τους επενδυτές στον τουρισμό. Και θέλω να δώσουμε προσοχή στο υψηλά καταρτισμένο εργασιακό δυναμικό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το 2016 363.000 άνθρωποι ε, εργάζονταν ε, σε θέσεις απασχόλησης που έχουν έμεση σχέση με το τουρισμό. Σε κάθε περίπτωση περιοχές αυτές, αναλόγως με το αν είναι χειμερινά ή θερινά, ε, χειμερινή ή θερινή τουριστική προορισμή, έχουμε υψηλότερη απασχόληση αναλόγως την αντίστοιχη εποχή του χρόνου. Σημαντικό είναι να δημιουργηθούν και είναι πρόθεση μας αυτή κέντρα κατάρτισης, εκπαίδευσης και επαγγελματικής ε, κατάρτισης έτσι ώστε να έχουμε ένα εργασιακό δυναμικό με υψηλά προσόντα. Όλα αυτά θα συμβάλλουν και στην προσέλκυση επενδύσεων. Το Υπουργείο Τουρισμού ε, ουσιαστικά χαρτογραφεί τις πιο πρόσφατες τάσεις για να καταλήξει σε απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο οι χρήστες, οι δημόσιες αρχές ε, ο ιδιωτικό τομέα θα ε, μπορούν να ε, βασίζονται στα στοιχεία του Υπουργείου για να χαράξουν πολιτική και στρατηγική. Είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα αυτή, όπου, την οποία θα τροφοδοτούμε με διάφορα στοιχεία. Από την 1η Ιανουαρίου του 2018 η Βουλγαρία θα έχει την Προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βασική προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της συνοχής και η προώθηση του τουρισμού. Το Υπουργείο Τουρισμού διοργανώνει δύο βασικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της Βουλγαρικής Προεδρίας, διάσκεψη υπουργική υψηλού επίπεδου για τον τουρισμό και την οικονομική ανάπτυξη το Φεβρουάριο και Διεθνές Φόρουμ για τον τουρισμό και την ενέργεια τον Μάιο. Θα αναλυθούν διάφορες πτυχές του τουρισμού πολύ σημαντικέ. Το 2018 επίση στη Βουλγαρία θα γίνει το ετήσιο φόρουμ τον Οκτώβριο του 2018 στη Σόφια για τη στρατηγική του Δούναβη με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στον τουρισμό, την οικονομική ανάπτυξη και την ενίσχυση τη συνοχή. Θέλω να σα ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, διότι διοργανώσατε αυτή τη σημαντική εκδήλωση, διότι μα δίνετε την ευκαιρία να συζητήσουμε για την προσέλκυση επενδύσεων, για τη δημιουργία φιλικού κλίματο προ τι επιχειρήσει επιχειρήσεις. Όλα αυτά θα τα δούμε και στο Συμβούλιο. Σε κάθε περίπτωση εμείς είμαστε δεσμευμένοι και προσιλωμένοι στο στόχο μας ο τουρισμός να γίνει πιο αηφόρος. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας. Ο Πρόεδρος και εγώ σας ευχαριστώ και ναι θα σας χρειαστούμε πολύ όταν η Βουλγαρία θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πράγματι ελπίζουμε ότι θα δοθεί υψηλή προτεραιότητα στο ε, τουρισμό, στο εξάμεινο της Προεδρίας σας. Ο κύριος Φρανσίσκο Μιγιάν συνάδελφός μου. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι Ευρωβουλευτής και συμπρόεδρος της Διακομματικής Ομάδας για την Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Τουρισμού, την Ανάπτυξη της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, δρόμο, τον δρόμο του Αγίου Ιακώβου, της Κομποστέλα και άλλων πολιτιστικών διαδρομών και επίσης ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε δύο πολύ σημαντικές πλατφόρμες. Έχουμε καταρχήν την επίσημη επιτροπή που είναι η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού που συνδέει τον τουρισμό με τις μεταφορές και έχουμε και ένα κίνημα με πάνω από 100 συναδέλφους μέλη ευρωβουλευτές που συμμετέχουν σε αυτή τη διακομματική ομάδα για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τουρισμού. Ο κύριος Φρανσίσκο Μιγιάν είναι συμπρόεδρος ε, της διακομματικής αυτής ομάδας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, εγώ θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα, οπότε βάλτε τα ακουστικά σας γιατί θα μιλήσω ισπανικά. Κύριε Αντιπρόεδρε Θελβέη, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι, εξοχότητες, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν ε, σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε και να ευχαριστήσω θερμότατα τον πρόεδρο Ταγιάννη για την πολύ επίκαιρη και εύστοχη αυτή πρωτοβουλία να συγκαλέσει αυτή τη διάσκεψη υψηλού επίπεδου για τον τουρισμό που συμπίπτει μάλιστα με την Παγκόσμια ημέρα του τουρισμού. Πρόκειται για μια πολύ εύστοχη πρωτοβουλία, γιατί όπως είπαμε ο τουρισμός αντιπροσωπεύει το 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, απασχολεί περίπου 17 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες και δυστυχώς το τελευταίο καιρό ο βάναυσος και στιγνός, η βάναυση και στιγνή τρομοκρατία έπληξε πολύ φημισμένες περιοχές του ευρωπαϊκού τουρισμού και μεγάλες πρωτεύουσες που τους τελευταίους μήνες ε, το Παρίσι, Βρυξέλλες, Βερολίνο, Νίκαια, Λονδίνο, Βαρκελόνη είναι από τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις που παρόλο που δέχονταν μεγάλο αριθμό τουρισμού πρόσφατα επλήγησαν από την ε, τρομοκρατική βαναυσότητα. Επίσης, είναι σημαντικό και συμβολικό που σήμερα από το οίκο των Ευρωπαίων πολιτών να διατρανώσουμε την εκτίμησή μας και την ε, μεγάλη αναγνώριση του τουρισμού στρατηγικού κλάδου, του τουρισμού και των τουριστών. Όπω αναφέρατε, κύριε Πρόεδρε, είμαι συμπρόεδρε τη Διακομματική Ομάδα για την Ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Τουρισμού, των Πολιτιστικών Κληρονομιών, των Δρόμων του Σατιάγκο, του Αγίου Ιακώβου και άλλων πολιτιστικών διαδρομών. Ω συμπρόεδρο λοιπόν αυτή τη Διακομματική Ομάδα, δεν θα σα εκπλήξει που θα μιλήσω για τη σημασία των ευρωπαϊκών πολιτιστικών διαδρομών που αναγνωρίζεται και από το Συμβούλιο τη Ευρώπη και που το 2017 συμπληρώνει 30 ετία. Μάλιστα είναι πάνω από 30 οι αναγνωρισμένες και επιστοποιημένε από το Συμβούλιο της Ευρώπης πολιτιστικές διαδρομές. Μερικέ από αυτές είναι οι δρόμοι του Αγίου Ιακώβου τη Κομποστέλα. Εγώ είμαι από τη Γαλλική, οπότε γνωρίζω αυτούς τους δρόμους, αυτές τις διαδρομές και για αυτές τις διαδρομές ε, που αναγνωρίστηκαν το 1997, ήταν οι πρώτες πολιτιστικές διαδρομές που αναγνωρίστηκαν. Θα σας μιλήσει εκτενέστερα αργότερα η Διευθύντρια του Τουρισμού της Γαλλικίας. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρουσιάσω κάποιες πτυχές που κατά τη γνώμη είναι πιο σημαντικές και αφορούν αυτές τις ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές. Καταρχήν, είναι πρώτη τάξη ε, τουριστικό αξιοθέατο οι διαδρομέ αυτέ, γιατί αναδεικνύουν σημαντικά στοιχεία τη ευρωπαϊκή ιστορία και τέχνη. Γιατί όλο και περισσότεροι τουρίστε ενδιαφέρονται για τον πολιτιστικό τουρισμό, όπω είπε και η Επίτροπο. Και από αυτή την άποψη, το 2018, που θα έχουμε το Ευρωπαϊκό Έτος Τουρισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Γνωρίζω ότι στη μεγάλη αυτή χώρα υπάρχει μεγάλο ζωηρό ενδιαφέρον για τον ευρωπαϊκό πολιτιστικό τουρισμό. Οπότε οι πολιτιστικές διαδρομές είναι σημαντικός ε, παράγοντας οικονομικής τόνωσης για τόπους και περιφέρειες που δεν εμπίπτουν στα κλασικά κυκλώματα ήλιου και παραλίας ή δεν είναι οι μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ή οι μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις. Έχουν όμως πολύ θετικό αντίκτυπο για την ύπεθρο, συμβάλλουν στην ανάπτυξη, ε, αποτρέπουν την έξοδο από τι πόλεις αυτές και επίσης δίνουν και απασχόληση στους νέου. Συμβάλλουν μάλιστα στη διαφύλαξη της ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς που με το πέρασμα του χρόνου διαβρώνεται. Αναβαθμίζουν κτίρια, ε, αρχιτεκτονικά μνημεία και εμφυσούν νέα πνοή σε όλα αυτά τα μνημεία. Και έχουμε και ένα πολύ πολιτικό επιπλέον ρόλο για τον οποίο είναι αξιόλογες αυτές οι πολιτιστικές διαδρομές. Οι διαδρομές αυτές αναδεικνύουν τους δεσμούς μεταξύ των Ευρωπαίων και αυτό το ε, κοινό ε, πολιτιστικό και ιστορικό υπόστρωμα που αποτέλεσε το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και από αυτή την άποψη για έναν Ευρωβουλευτή όπως εγώ είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βοηθήσουμε τις διαδρομές αυτές τις πολιτιστικές και να διευκολύνουμε τις ε, χρηματοδοτήσεις ε, και από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από το Κόσμε μπορούμε να βρούμε κονδύλια για τις ε, διαδρομές αυτές. Και μάλιστα το 2018 που θα είναι έτος της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα πρέπει να κάνουμε μια επιπλέον προσπάθεια να βοηθήσουμε αυτές τις περιοχές που συγκεντρώνουν τόσα πολλά στοιχεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και από το σχέδιο Juncker, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε τέτοιε διαδρομέ. Για παράδειγμα, στην Ισπανία, ο ε, κρατικός φορέας δανεισμού σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει προβλέψει μια γραμμή πιστοτική για να ε, προωθήσει ε, σχέδια ενεργειακής απόδοσης για τον τομέα τον ξενοδοχειακό. Ο πολιτικός τουρισμός λοιπόν έχει λαμπρό μέλλον και πολύ μεγάλη σημασία. Και σημασία έχει όχι μόνο για τις περιοχές που διασχίζουν αυτές οι διαδρομές, αλλά για το σύνολο του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Φρανσίσκο, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Όπως είπα και προηγουμένως, χρειαζόμαστε πραγματικά τον ευρύτερο συνασπισμό ε, των μεγαλύτερων ομάδων. Είχαμε τον κύριο Μιγιάν από το ΕΛΚ, τώρα θα έχουμε τον καλό μου φίλο από του Σοσιαλιστέ και δημοκράτε τον κύριο Μιλτιάδη Κύρκο, που είναι Ευρωβουλευτής και μέλος Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. Μιλτιάδη, έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Dear friends, this Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, φίλο μου και πρόεδρο σήμερα για τις προσπάθειες που κατέβαλε ε, για τη σημερινή συνάντηση και να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο κύριο Ταγιάννη ο οποίος ε, μας βοήθησε να έχουμε αυτή την θαυμάσια συνεδρίαση. Ευχαριστώ την κυρία Καφαντάρη από την ελληνική κυβέρνηση. Εμείς είμαστε στην αντιπολίτευση, αλλά όπως είπε και ο κύριος Αγιάννη, υπάρχουν πολλά θέματα που είναι πέρα από τα κόμματα. Επενδύσεις λοιπόν, όλοι μιλάνε για επενδύσεις. Πώς μπορούμε να προσελκύσουμε νέες επενδύσεις, μπορούμε να το επιτύχουμε ε, ευαισθητοποιώντας περισσότερο και αυτό που ενδιαφέρει είναι όχι μόνο πώς να έχει κανείς πρόσβαση στο ΕΦΣΙ, αλλά πώς να συνδυάσει αυτή την οικονομική εγγύηση με άλλα ε, χρηματοπιστωτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που αποκαλείται blending, την ανάμειξη των διαφόρων εργαλείων. Ε, γιατί αυτό θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Όσον αφορά τις τομεακές ανισορροπίες, χαιρόμαστε που η Επιτροπή του Κοινοβουλίου κατόρθωσε τον τουρισμό να τον βάλει σε πρώτη προτεραιότητα στον κανονισμό για το ΕΦΣΥ. Και ελπίζουμε αυτό να σημάνει πολλά νέα προγράμματα για τον τουριστικό τομέα. Ως προς την γεωγραφική ανισορροπία, η γεωγραφική κάλυψη που προσφέρει ο ΕΦΣΥ θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω κυρίως σε λιγότερο εξόχως απομακρυσμένες περιοχές, σε μικρά νησιά όπως ε, στην κοιλάδα το Χελόου, γιατί πρέπει τέτοιου είδου ε, τοποθεσίες να ληφθούν ιδιαίτερα υπόσψη. Αγαπητοί φίλοι, το πρόγραμμα ΕΦΣΥ, στρατηγικό επενδύσεις ε, στρατηγικού σχεδιασμού δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα πάντα, για να, πάντα για να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη και την ανταγωνιστικότητα. Όσον αφορά την Ελλάδα, πρέπει να ξεπεράσουμε τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, γενικότερα ε, να υπάρχει μια σταθερότητα, να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες όσον αφορά την ε, γραφειοκρατία, γιατί όλα αυτά ε, διαταράσουν τα επενδυτικά προγράμματα. Ο αντιπρόεδρος κ. Κατάινεν πριν από ένα χρόνο μίλησε για τη δυνατότητα άλλες χώρες να αντιγράψουν την τουριστική πλατφόρμα που ήδη υπάρχει στην Κύπρο ε, που δίνει τη δυνατότητα μικρές και μεγάλες επενδύσεις ε, να συγκεντρώνονται. Μία πλατφόρμα που συγκεντρώνει πρωτοβουλίες και ευκαιρίες, διότι η συμβολή του δημόσιου τομέα είναι απολύτως απαραίτητη για τον συντονισμό των αναγκών. Πρέπει να υπάρχει μία πλατφόρμα που να προσφέρει χρηματοψηφιακή αλλά και τεχνική αρρωγή πρόσφατο παράδειγμα που δείχνει γιατί η Ελλάδα, ενώ έχει τεράστιες δυνατότητες για τουριστικές επενδύσεις, δεν είναι πρώτη προτεραιότητα. Πάμε στην ακτογραμμή μας ε, και στη δυνατότητα των νησιών να συνδέονται μεταξύ τους. Πολλές φορές όμως τα νησιά δεν συνδέονται μεταξύ τους. Πρέπει κανείς να επιστρέψει στην ε, υπηρετική Ελλάδα και να ξαναπάει σε επόμενο νησί. Ε, εγκρίθηκε ένα πρόγραμμα για τα, τα αεροπλάνα, υδροπλάνα με συγχωρείτε, η κυβέρνηση λοιπόν όμως ε, έχει προβλέψει ένα νέο νόμο που απαγορεύει τις ε, επενδύσεις στα υδροπλάνα και έτσι το πρόγραμμα κυρώθηκε. Θα ήθελα να επισημάνω λοιπόν ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό πλαίσιο. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να είναι προβλέψιμο, να ευαισθητοποιεί μακροχρόνιες επενδύσεις ε, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και πέρα από τα χρηματοψηφιακά εργαλεία, είναι σημαντικό να στηριχτούν οι χώρες έτσι ώστε να συγκλίνουν γιατί δεν είναι δίκαιο να μιλάει κανείς για ίσες ευκαιρίες ε, στις ε, επενδύσεις όταν σε κάποιες χώρες η δικαιοσύνη αποδίδεται σε δύο ή πέντε χρόνια και σε άλλες σε 15. Εμείς είμαστε ακράδαντα πεπισμένοι ότι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση είναι πολύ πιο βαθιά από απλά και μόνο τα οικονομικά εργαλεία. Και να πω ότι παρότι το πρόγραμμα Juncker είναι πολύ πετυχημένο, δεν πρέπει να αντικαθιστά τα ταμεία συνοχής καθοριστικής σημασίας για τις οικονομίες μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αποβλέπει στην σύγκληση και το κλείσιμο του χάσματος ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Ε, πρόεδρος, ε, χαίρομαι που μπορώ να σας πω ότι το τουριστικό λόμπι της Ελλάδας είναι όλο και πιο δυνατό. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα έχουμε ένα νέο διευθυντή που θα είναι Έλληνας και θέλουμε να πιστεύουμε ότι από κοινού θα στηρίξετε τον τουρισμό. Επόμενος είναι ο κύριος Μάσιο Φαΐλια, πολύ καλός φίλος μου, ο οποίος ε, υπηρέτησε τον τουρισμό στην κυβέρνηση της Βραζιλίας κατά το παρελθόν. Είναι από τη Μαδρίτη, είναι εκτελεστικός διευθυντής ε, του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών. Και όπως είπα, σε προηγούμενη παρέμβασή μου, κατά τους επόμενους μήνες, δεν ξέρω ακριβώς πότε, αλλά θα έχουμε μια επίσημη συμφωνία ανάμεσα σε αυτόν τον οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών και, του, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ελπίζω θα είναι ένα νέο βήμα για να ε, στηριχθούν οι ευρωπαϊκοί φορείς που ασχολούνται με τον τουρισμό. Έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αγαπητοί πρέσβεις, διακεκριμένοι προσκεκλημένοι. Εκ μέρους του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, της Ειδικής Υπηρεσίας των Εθνών για τον Τουρισμό, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μας εκτίμηση στον Πρόεδρο Αντώνιο Ταγιάννη για τη διοργάνωση αυτής της, της εκδήλωσης υψηλού επίπεδου και για την πρόσκληση που μας απίφθενε σε αυτή την πολύ σημαντική μέρα για εμάς και για την παγκόσμια τουριστική κοινότητα. Από τη στιγμή που σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Το 2017 είναι μια σημαντική χρονιά για όλους μας, γιατί γιορτάζουμε και το ε, έτος ε, για την αηφόρο τουριστική ανάπτυξη, για τον αηφόρο τουρισμό και ανάπτυξη. Είναι ένα έτος που είναι ευκαιρία για να ε, ενισχύσουμε την συνέστηση του κοινού, να κινητοποιήσουμε τους εταίρους, τα εμπλεκόμενα μέρη, έτσι ώστε ο τουρισμός να λειτουργήσει καταλυτικά για θετικές αλλαγές και στις ανεπτυγμένες και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Κυρίες και κύριοι, παρά τις πολλές πολιτικές και οικονομικές προκλήσεις σε πολλά μέρη του κόσμου και στην Ευρώπη, ο τουρισμός το μόνο που κάνει είναι να αυξάνεται. Και κυρίως στην Ευρώπη, που είναι η πιο συχνά επισκεπτόμενη περιοχή του κόσμου. Όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οθέτησε την ανακοίνωσή της, Ευρώπη υπαριθμών ένα τουριστικός προορισμός παγκοσμίω, ένα νέο πλαίσιο, οι αφήξει στην Ευρώπη έφτασαν στα 400 τόσα εκατομμύρια, ενώ πέρσι έφτασαν οι αφήξεις στα πάνω από 600 τόσα εκατομμύρια, 26% αύξηση μέσα σε 6 χρόνια, κάτι το οποίο είναι το 50% όλων των διεθνών αφήξεων. Τους πρώτους 6 μήνες του 2017 στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημειώθηκε αύξηση κατά 8% των διεθνών αφήξεων και αυτό είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτές οι θετικές τάσεις αναμένεται να συνεχιστούν. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο τουρισμός είναι βασικός κινητήριος μοχλός για την ανάπτυξη και ε, ε, βασικός μοχλός για τη δημιουργία άμεσων και ε, άμεσος και έμεσος μοχλός για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνει ευκαιρίες σε νέους, δίνει ευκαιρίες για επενδύσεις και σε παραδοσιακές και σε μη παραδοσιακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις, δίνει ευκαιρίες στους πιο ταλαντούχους επιχειρηματίες. Όλα αυτά είναι βασικά χαρακτηριστικά των χωρών μας. Η Ευρώπη έχει το, τους φυσικούς, πολιτιστικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς ε, πόρους για να παραμείνει τουριστικούς προορισμούς τα επόμενα χρόνια, βασικό και μόνιμο σημείο αναφοράς. Χρειάζεται ο τουρισμός πολυκλαδική, διατομεακή προσέγγιση, στενή συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Υπ' αυτή την ενέα. Στην τελευταία μας συνεδρίαση, η συνεδρίαση των ανώτατων τουριστικών αρχών των χωρών του G20 με στήριξη του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού, στην οποία παρέστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή, ε, υιοθετήθηκε μια διακήρυξη για τη δυνατότητα του τουρισμού να ενισχύσει την ανάπτυξη και την ε, δημιουργία θέσεων απασχόλησης και αναγνωρίστηκε επισήμως ότι είναι πολύ σημαντικό να ε, παρακολουθούμε την αγορά εργασίας στην τουριστική, την αποτελεσματική αξιοποίηση εργασιακού δυναμικού με προσόντα, με δεξιότητες και ε, να ε, αναγνωρίσουμε ότι ο τουρισμός ενισχύει την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Επίσης, στη διακήρυξη ε, συμπεριλήφθηκε η ανάγκη να γίνει περαιτέρω έρευνα για να δούμε ποια είναι τα κενά που χρειάζεται να καλυφθούν ανάμεσα στην εκπαίδευση από τη μία και τις, αυτό που ζητάει η αγορά από την άλλη. Τρίτον, Σημαντικό είναι να ενισχυθούν οι επενδύσεις στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο τομέα του τουρισμού και τέταρτον θα πρέπει να απεικονίζονται με μεγαλύτερη ορατότητα τα ωφέλη των δουλειών, των εργασιών στον τομέα του τουρισμού για να προσελκύσουμε ταλέντα στο χώρο μας. Κυρίες και κύριοι, Πέρσι, ένα δις 200 εκατομμύρια ταξιδιώτες διέσχισαν τα σύνορα της χώρας τους. Μέχρι το 2030 αυτό το 1,2 δις θα γίνει 1,8 δις. 1,8 δις ευκαιρίες λοιπόν να αλλάξει η ζωή προς το καλύτερο, να προστατευτεί ο πλανήτης και να εξασφαλίσουμε ανάπτυξη για όλους και δημιουργία θέσεων απασχόλησης για όλους. Inclusive. Πώς μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό για να συμβάλλουμε στην, στο θεματολόγιο για την αηφαρό ανάπτυξη. Αυτή είναι η ερώτηση που πρέπει να απευθύνουμε κάθε μέρα, κάθε χρόνο στους εαυτούς μας και πόσο μάλλον φέτος που είναι το ευρωπαϊκό έτος για τον αηφόρο τουρισμό και την ανάπτυξη. Ένα έτος που ε, εστιάζει την προσοχή του στον τουρισμό και στην ικανότητά του να ενισχύσει την ανάπτυξη και την επίτευξη των στόχων ε, της χιλιετίας και των ε, στόχων της η φόρα ανάπτυξη των 17 που καθορίστηκαν στη Σύνοδο των Παρισίων. Θα πρέπει να προχωρήσουμε προ μια πραγματικά πράσινη οικονομία. Η ανάπτυξη να αποσυνδεθεί από το πλήγμα στο περιβάλλον και να αποσυνδεθεί από την εξάρτηση των φυσικών πόρων. Καινοτομία, επένδυση, ε, προσοντούχο εργασιακό δυναμικό χρειάζεται θα πρέπει να μετρηθεί ο αντίκτυπος της τουριστικής έλευσης με ακρίβεια για να διαχειριστούμε καλύτερα τους κλάδους και τους τουριστικούς προορισμούς. Θα πρέπει να προωθήσουμε την προσβασιμότητα σε όλους, να εντάξουμε, να εμπλέξουμε τις τοπικές κοινότητες, να εξασφαλίσουμε ότι τα ωφέλη που δρέπει ο τομέας θα φτάσουν στην τοπική κοινωνία, θα τα δρέψει και εκείνη. Και τέλος θα προστατέψουμε, να προστατέψουμε τους αδύναμους και αυτούς που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση τι πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτή η απόσταση πρέπει να καλυφθεί. Είμαστε υπεύθυνοι για το 5% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά για να μειώσουμε αυτό το ποσοστό. Ένας τουριστικός τομέας με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, με χαμηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρωπα θα πρέπει για να το πετύχουμε να δεσμευθούν ε, και οι αερομεταφορεί και οι αεροπορικές υποδομές και τα υπόλοιπα συστήματα μεταφορών και τα ξενοδοχεία ξενοδοχεία και υπηρεσίε απανταχού, ε, ξενοδοχειακέ και εστίασης και άλλες. Μας ενδιαφέρουν ε, οι ενεργειακές λύσει στα ξενοδοχεία, τα ενεργειακά ξενοδοχεία με σχεδόν μηδέν ενεργειακό ε, αποτέλεσμα στο ενεργειακό ισοζύγιο και εμπλοκή και ενεργή συμμετοχή των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ξέρουμε ότι ο τουρισμός συμβάλλει άμεσα και έμεσα στο 10% του παγκοσμίου ΑΕΠ. Μία στις 10 δουλειέ έχουν να κάνουν ε, με το τουρισμό. 7% του παγκοσμίου εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών έχει να κάνει με το τουρισμό. Είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό για την ευρωπαϊκή οικονομία και για τον τρόπο ζωής των Ευρωπαίων αφού θα φτάσουμε 1,8 δις αφήξεις από το εξωτερικό το 2030, χώρια τα ταξίδια και τη τουριστική δραστηριότητα εντός των σύνορων κάθε χώρας ε, δεν είναι το πρόβλημα η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη είναι το εργαλείο για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Ο τρόπος που θα προχωρήσουμε προς τα εμπρός με καινοτομία, με ανάπτυξη των τεχνολογιών, με επενδύσεις, με το να διασφαλίζουμε ότι γίνεται σωστή διαχείριση του τουρισμού και είναι αυτός βιώσιμος, αηφόρος σε όλες τις διαστάσεις του, ε, τούτων λεχθέντων δεν τίθεται το ρέμα του αν θα πρέπει να αναπτυχθούμε, αλλά το πώς θα πρέπει να αναπτυχθούμε και άρα ως ε, Ηνωμένα Έθνη θέλουμε, ως Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού θέλουμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και να στηρίξουμε τις πρωτοβουλίε σας. Έτσι ώστε ο τουρισμός να καταστεί μια πραγματικά δύναμη μετασχηματισμού, δύναμη του καλού ε, που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αυτό που γίνεται στην Ευρώπη εμπνέει και τον υπόλοιπο κόσμο. Ε, ε, ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στο έργο όλων σας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε αγαπητέ Μάρσιο, κύριε εκτελεστική διευθυντά της Παγκόσμιας Οργάνωσης Τουρισμού και μεταφέρετε θερμές ευχές προς συναδέλφους σας από εμά στον κύριο Σάλαμπρη, τον Ζόλταν Πίτερ και τους υπόλοιπους. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Μάουρο Παρολίνη Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης της ε, Περιφέρειας της Λομβαρδίας. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Καλημέρα, εγώ θα μιλήσω Ιταλικά. Η περιοχή της Λομβαρδίας είναι μια περιοχή που είναι γνωστή κυρίως ε, για το σύγχρονο σχεδιασμό για τις υπηρεσίες ε, που προσφέρονται στον τριτογενή τομέα. Τα τελευταία χρόνια έγινε μία από τις ε, πιο σημαντικές ε, τουριστικές περιοχές της Ιταλίας και έχει ένα χαρακτηριστικό. Δεν έχει περιορισμένη προσφορά. Οι πόλεις δεν προσφέρουν μόνο τουρισμό, ούτε μόνο την λίμνη και τα βουνά. Έχει μία βεντάλια προσφορών στην πραγματικότητα λοιπόν ο τουρισμός στη Λομβαρδία έχει, αποτελείται από πολλές μικρές επιχειρήσεις. Υπάρχει κάποιος κατακαιρματισμός. Οι οποίες μικρές αυτές επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να συγκεντρώσουν πολλούς επιχειρηματίες και να αποδεικνύουν δυναμισμό. Όμως ε, αυτό σημαίνει ότι πρέπει και αυτοί κάπως να στηριχθούν σε, παγκόσμιο, σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Η Λομβαρδία έχει τουρισμό ο οποίος ε, τα τελευταία τρία χρόνια χαρακτηρίζεται από το εξής. Αφενός, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δώσουμε μία φωνή στην τοπική πραγματικότητα, δηλαδή αυτό που δεν μπορεί ο καθένας να το κάνει μόνος του, να το κάνουν πολύ περισσότεροι σε περιφερειακό επίπεδο. Άρα μας ενδιαφέρει να ξεπεραστεί ο κατακαιρματισμός μέσα από μία σειρά εργαλείων που επιτρέπουν την χρήση νέων εργαλείων και με τον τρόπο αυτό να προσαρμόζεται κανείς πιο συγκεντρωμένα. Υπάρχει όμως από την άλλη και η αναγκαιότητα να μην υπάρχει ομοιογενοποίηση γιατί η προσφορά στην Ιταλία αλλά και γενικότερα στην Ευρώπη ακριβώς αυτό είναι, είναι η διαφοροποίηση, η βεντάλια που σας είπα προηγουμένως. Έχουμε πάρα πολλές ε, ε, προσφορές, πολλές δυνατότητες να επισκεφτεί κανείς ως τουρίστας Άρα δηλαδή έχουμε δύο γεγονότα. Την ε, πραγματικότητα, τον κατακαιρματισμό αφενός και αφετέρου το να προβάλλουμε αυτή την ε, διαφοροποίηση. Είναι δύο στοιχεία που μοιάζουν ε, ότι δεν συνδέονται μεταξύ τους, αλλά δεν είναι αλήθεια εμείς μπορούμε να δώσουμε δυνατότητα στην τοπική κοινωνία να έχει πιο δυνατή φωνή. Και ως ε, εκ τούτου ε, θέλουμε να προβάλλουμε αυτές τις ε, διαφορές. Υπάρχει και κάτι άλλο. Η πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια στον τουρισμό είναι εξή. Έχουμε, έχει αυξηθεί κατά έξι φορές παραπάνω από μεσοσταθμική αύξηση του ΑΕΠ. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έχουν γίνει και πάρα πολλές ιδιωτικές επενδύσεις. Η περιοχή της ε, Λομβαρδίας ε, προσπάθησε να στηρίξει όλους αυτούς τους επενδυτές. Για πρώτη φορά μπορέσαμε και να εκμεταλλευτούμε τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτό λοιπόν οδήγησε σε περαιτέρω προσέλκυση επενδύσεων. Ως εκ τούτου, ο τουρισμός στη Λομπαρδία έχει αυξηθεί όχι μόνο αριθμητικά, αλλά και στην προστιθέμενη αξία και ως εκ τούτου και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ποιο είναι τώρα το καθοριστικό στοιχείο πέρα από αυτά που σας ανέφερα και πέρα από την ποιότητα των επενδύσεων, το γεγονός ότι ο τουρισμός είναι μια σχετική οικονομία, δηλαδή βασίζεται κυρίως στις δυνατότητες και στην εκπαίδευση των άμεσα ενδιαφερομένων. Εμείς λοιπόν έχουμε δώσει ιδιαίτερη σημασία στην διάχυση των αρμοδιοτήτων αλλά και σε μια τέτοια νοοτροπία που θα εκμεταλλεύεται αυτό που υπάρχει θέμα της εκπαίδευσης των επιχειρηματιών, αυτό είναι ένα θέμα καθοριστικής σημασίας. Και είναι αλήθεια ότι ο δικός μας ο στόχος είναι να γίνουμε η πρώτη τουριστική περιοχή της Ιταλίας. Αυτό βασίζεται ακριβώς σε αυτό που σας εξήγησα, δηλαδή στο να εκπαιδεύσουμε τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Τι ζητάμε από την Ευρώπη είναι να κάνει η Ευρώπη αυτό που λιγάκι κάνουμε και εμείς, δηλαδή να προβάλλει τις διαφορές, να συντονίσει τις προσπάθειες και να καταστήσει απέναντι ότι αυτό που δεν μπορεί να κάνει κανείς μόνος του μπορεί να το κάνουν περισσότεροι και όλοι μαζί. Διατηρείται βέβαια αυτονομία και μέσα από τη συνεργασία. Στην ε, δική μας περίπτωση έχουμε τις περιφέρειες που συνεργάζονται, στην Ευρώπη θα έχουμε τα κράτη που θα συνεργάζονται με τον τρόπο αυτό η Ευρώπη θα μπορεί να έχει μια ξεκάθαρη τουριστική πολιτική. Ως εκ τούτου ζητάμε από την Ευρώπη να μας βοηθήσει στο συντονισμό η ε, Ευρώπη να εμφανίζεται με πιο ηχηρή φωνή σε παγκόσμιες αγορές και να ε, εκμεταλλεύεται αυτό που χαρακτηρίζει την κάθε χώρα ξεχωριστά. Να υπάρξουν κονδύλια που σήμερα αυτά είναι περιορισμένα, είτε άμεσε ενισχύσει, είτε αυτά που χορηγούνται μέσα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που πρέπει να αυξηθούν, αλλά κυρίω πρέπει να διατίθενται στου άμεσα ενδιαφερόμενου με προσαρμογή στον οικονομικό αυτό τομέα που σας λέω αποτελείται από πολλούς μικρούς παράγοντες. Αν η οικονομική βοήθεια δεν ε, συμβάλλει στο να βελτιωθεί η προβολή και η ε, άμεση βοήθεια στις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτό θα είναι ένα πλήγμα. Θεωρώ ότι εμείς μπορούμε πλέον να περιμένουμε μια Ευρώπη που θα είναι όλο και πιο παρούσα ακόμα και στον τομέα του τουρισμού. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, χίλια ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ. Επόμενος ομιλητής μας είναι ο κύριος Κλάους Βίγκλερ που είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Εθνικών Ενώσεων Ξενοδοχείας Εστίασης και Αναψυχής της HOTREC. Ξέρετε ότι η είναι από τους βασικούς ενδιαφερόμενους και από τους πιο δραστήριους ε, και συνεργάζεται στενά με τους ευρωβουλευτές. Η Ευρωπαϊκή αυτή οργάνωση πάντα προσκαλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσμικό όργανο κάθε φορά που οργανώνει εκδηλώσεις ή διασκέψεις. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν η συνεργασία HOTREC και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κυρία Πρόεδρε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την εισαγωγή σας. Κύριε Επίτροπη, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κύριε και κύριοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι μαζί σα για να εορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού και μετά όλε τι ομιλίε που ακούσαμε και όπω είπε και ο Πρόεδρο Ταγιάννη, ο τουρισμό βρίσκεται όντω στην καρδιά τη Ευρωπαϊκή Οικονομία. Ακούσαμε πολλά στοιχεία για τον τουρισμό σήμερα, αλλά ας μην ξεχνάμε και τις προκλήσεις, ε, κυρίως ε, για το κλάδο των ξενοδοχείων, που απασχολεί το 80% των ε, θέσεων απασχόλησης, αντιπροσωπεύει το 80% των θέσεων απασχόλησης του κλάδου τουρισμού. Και αν θέλουμε να επωφεληθούμε ε, πλήρως από βιώσιμο και υγιή κλάδο θα πρέπει να δημιουργήσουν τα θεσμικά όργανα ένα πλαίσιο πολιτικής που θα προωθεί και την επιχειρηματικότητα και θα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 99% των ε, ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων στον τουρισμό είναι μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οπότε θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα εργαλεία, τους μηχανισμούς και τους στόχους και να μην μιλούμε μόνο για τεχνολογική επανάσταση και ψηφιοποίηση. Αυτό θα έρθει αργότερα. να δούμε ποιοι είναι οι δικοί μας στόχοι και ποιους στόχους θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε εδώ. Καταρχήν, φορολογία. Ε, η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα του τουρισμού σχετίζεται άμεσα με ε, τις επενδύσεις που γίνονται και το πόσο αποδοτικές είναι αυτές. Και μια και ο τουρισμός ε, διεθνώς αυξάνει ε, παντού, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικό να έχουμε χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχουμε τουριστικά προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικές, ειδικούς φόρους που έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην τιμή, ενώ ε, το εισόδημα, τα κέρδη που αποκομίζονται δεν επανεπενδύονται στις υποδομές. Και μάλιστα η Χοτρέκ και οι ενώσεις χρειάζονται μόνιμη εφαρμογή χαμηλών φορολογικών συντελεστών για την ξενοδοχεία, εστίαση και αναψυχή, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του κλάδου στο παγκόσμιο στην παγκόσμια αγορά και να παραμείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτο υπαριθμό τουριστικό προορισμό στον κόσμο. Επίση, ε, ο νόμο ε, για την σήμαση. Η εποχιακή διάρθρωση του τουρισμού σημαίνει ότι ε, δεν μπορούν όλε οι εταιρείε να προσφέρουν μόνιμες συμβάσεις απασχόλησης, ενώ επίσης οι πελάτες περιμένουν να είναι μονίμως στο απίκο και διαθέσιμες οι τουριστικές υπηρεσίες όλο το 24ωρο και όλο το χρόνο. Οπότε κάποιες ελαστικές ρυθμίσεις απασχόλησης είναι σημαντικές για τον κλάδο αυτό. Νέο κόστος και διοικητικό άχθος, όπως είναι υποχρεωτικές ε, ε, άδειε που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ανέφικτε για μας λόγω των χαρακτηριστικών ε, του κλάδου και των απαιτήσεων των πελατών. Οπότε ο συνδυασμό οικογενειακού και επαγγελματικού κλάδου μπορεί να επιτευχθεί, με άλλου τρόπου, με καλύτερη λειτουργία των βρεφονιπιακών σταθμών, για παράδειγμα, με ευρύτερο ωράριο. Επίση, ο μέσο των ξενοδοχείων αντιμετωπίζει τεράστια έλλειψη δεξιοτήτων. Και έχουμε πολλά, ε, πολλές κενές θέσεις, πολύ περισσότερες στον κλάδο αυτό από ότι στο, την υπόλοιπη οικονομία. Ενώ θέλουμε να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση, δεν βρίσκουμε την ειδίκευση και τη δεξιότητα που χρειαζόμαστε ή τι απαραίτητε καταρτήσει για την ψηφιοποίηση που απαιτεί ε, ευρωπαϊκά κονδύλικα. Οπότε θέλουμε και καλύτερα προγράμματα για, για την άσκηση και την κατάρτιση. Αυτά θα πρέπει να επεκταθούν και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να διευκολύνουν τη μετάβαση από τις σπουδέ ε, στην απασχόληση με αύξηση των δεξιοτήτων. Θα μπορούσα ώρες ολόκληρες να σας ε, μιλάω για το τι χρειάζονται για να βελτιωθεί ο τουρισμός, αλλά προς το παρόν σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω σε μια καρποφόρο συζήτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω ότι η Ένωση σα, η Χοτρέκ, θα συνεχίζει να στηρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα στηρίζει τη Χοτρέκ και τα μέλη τη τι Εθνικέ ενώσει, δηλαδή ξενοδοχεία, εστίαση και αναψυχής. Επόμενο ομιλητή, είναι ο κ. Πίτερ Ντεβίλτε, που είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ταξιδιών, της ETC, που είναι από τους σημαντικότερου και πιο δημοφιλείς ε, ενδιαφερομένους ε, ε, μια οργάνωση που έχει την έδρα της Βρυξέλλες. Άρα ο Πίτερ βρίσκεται στην πατρίδα του, είναι από τη Φλάνδρα και θα μας δώσει πληροφορίες για τα μελλοντικά σχέδια της ε, οργάνωσής του της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής Ταξιδιών. Παρακαλώ, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι εξοχότητες, είναι καλό που μιλάει για σήμερα το απόγευμα κάπως αργά γιατί οι προλαλήσαντες με έχουν καλύψει σε μεγάλο βαθμό, γι' αυτό θα εστιαστώ στα βασικά. Όταν διάβασα την πρόσκληση για αυτό το φόρουμ, είδα ότι γίνεται λόγος για τα διοικητικά εμπόδια και τη γραφειοκρατία. Και θεώρησα ότι με καλείται για να σχολιάσω και αυτό το ζήτημα, λόγω της ιδιότητάς μου. Κάποιος προσκεκλημένος μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας μίας ευρωπαϊκής υπηρεσίας τουρισμού. Και όταν το άκουσα δεν μπορώ να πω ότι πανικοβλήθηκα, αλλά μπορώ να πω ότι δεν νομίζω ότι είναι πολύ καλή ιδέα. Αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών κρατών μελών, όπω το κάνουμε άλλωστε υπό την αιγίδα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών, μέλη τη οποία είναι 33 χώρε τη Ευρώπη, είναι και το καλύτερο. Η Επιτροπή επέλεξε να δώσει περισσότερες δυνατότητες σε αυτή τη μορφή συνεργασίας και είναι μια σόφρονα ε, μια πολύ σοφή απόφαση. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερε υπηρεσίε, αλλά περισσότερη συνεργασία, καλύτερη συνεργασία, πιο δημιουργική συνεργασία. Και ε, σε καιρού σαν του σημερινού, όπου έχουμε πολιτικές αναταραχές, όπου έχουμε προβλήματα ασφαλείας, αυτό χρειαζόμαστε περισσότερη και καλύτερη συνεργασία. Οι τουρίστε θα συνεχίσουν να εξερευνούν τι περιοχέ μα και οι προβλέψεις είναι πολύ θετικέ προβλέπεται αύξηση των αφήξεων κατά 3% ε, σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ταξιδιών και ε, οι ευρωπαϊκοί προορισμοί θα συνεχίσουν να ε, ε, αποτελούν ε, στόχο για τους τουρίστες για το 2017. Και αυτό φαίνεται από το δίκτυο εντυπώσεων που έχουμε για τα υπερατλαντικά ταξίδια, τα ταξίδια μακρινών αποστάσεων. Ωστόσο, ο ελέφαντας στο δωμάτιο είναι το θέμα των θεωρήσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει μερίδιο της αγοράς γιατί οι αναδυόμενες οικονομίες αναπτύσσονται πιο γρήγορα και περισσότερο. Σύμφωνα με την έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για το πόσο εύκολο είναι να έχει κανείς θεώρηση εισόδου, το καθεστώ στην Ευρώπη είναι και το πιο περιοριστικό. Η δημιουργία του χώρου Σέγγεν έχει συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση των ταξιδιών εντό Ευρώπη, αλλά έκανε και την Ήπειρό μα λιγότερο προσβάσιμη για ταξιδιώτε από, το, από τρίτες χώρες εκτός Ευρώπης. Οι πολίτε από τι περισσότερε χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται θεώρηση για να έρθουν στην Ευρώπη και οι κανόνε του Σέγγεν δεν είναι και οι μόνοι κανόνε που εφαρμόζονται. Έχουμε ε, πραγματικότητες εντός Σέγγεν, αλλά εντός Ευρώπης, ευρύτερε πέραν των χωρών Σέγγεν, αλλά μη Ευρωπαϊκή Ένωση, όλα αυτά με μεταβλητές γεωμετρίες, κάτι το οποίο περιπλέκει τα πράγματα για τους Κινέζους τουρίστες και για άλλους τουρίστες. Όλα αυτά ε, αποτελούν τροχοπέδι στην ανάπτυξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών έκανε μια μελέτη για το πόσο θα μπορούσαμε να διευκολύνουμε τις διαδικασίες και την κατάσταση για τις θεωρήσεις. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες αντιδράσεις για τις θεωρήσεις και ποιο αντίκτυπο θα έχει αυτό στην ευρωπαϊκή οικονομία. Αναλύσαμε 10 βασικές ε, αγορές προέλευσης τουριστών και τα ευρήματα πάντοτε επιβεβαιώνουν και τις προηγούμενες έρευνες. Όσο περισσότερο έχουμε απελευθέρωση του καθεστώτος, τόσο μεγαλύτερα θα είναι ε, τα οικονομικά ωφέλη. Αν ε, καταργήσουμε τις θεωρήσεις για τα για ταξιδιώτες από αυτές τις 10 αγορές θα έχουμε 84 εκατομμύρια περισσότερες αυξήσεις, περισσότερα δις δαπάνες στα πόσο ξοδεύει ο κάθε τουρίστας και πάρα ε, πολλές θέσεις απασχόλησης και τα νούμερα είναι πολύ συγκεκριμένα και μιλούν από μόνα τους. Θέλω λοιπόν να παρακινήσω όλους τους ηθήνοντες υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής να αξιοποιήσουν τα ερευνητικά δεδομένα που, στα οποία έχουμε καταλήξει εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών αλλά και στα άλλα θεσμικά όργανα. Και υπό αυτή την έννοια θα ήθελα, και από την που είμαι και από το Βέλγιο, δεν μπορώ να το πράξω και διαφορετικά, θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο Αναβράτσιτς, διότι αναφέρθηκε στην έρευνα ε, τη δική μας. Ε, και την έρευνα που έγινε στην πόλη της Μπρίζ στο Βέλγιο για τη στάση των κατοίκων ε, ως προς τον τουρισμό. Είναι μια μεθοδολογία που εξάγουμε σιγά σιγά και συνομιλούμε με άλλες περιοχές και πόλεις στην Ευρώπη που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Πιστεύουμε ότι όταν διαδίδεται η γνώση, όταν μοιραζόμαστε την πληροφορία, αυτό είναι το κλειδί για την επιτυχία στην Ευρώπη. Ενίσχυση συνεργασίας, ενίσχυση του διαμοιρασμού της γνώσης, αυτά θέλουμε να τονίσουμε σήμερα. Για ώρες θα μπορούσα να μιλάω όπως και όλοι ε, οι άλλοι ομιλητές, αλλά δεν θα ήταν αυτό δίκαιο για τους υπόλοιπους. Γι' αυτό και θα σταματήσω κάπου εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ναι, ξέχασα να το πω ότι θα έχετε, Πίτερ, συζήτηση εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα του μαζικού τουρισμού. Θα έχουμε ομιλητές από την Ιταλία, από τη Βαρκελόνη, από την Κροατία, θα ήταν ενδιαφέρον και εσείς να παραστείτε σε αυτή τη συζήτηση για το μαζικό τουρισμό και να μοιραστείτε μαζί μας πληροφορίες για την κατάσταση στην Πρίζ. Θα σας στείλω πρόσκληση για, αυτό το, για αυτή την εκδήλωση. Επόμενος ομιλητής είναι ο κ. Τζιανφράνκο Μπατίστη, πρόεδρος της Φεντέρ Τουρισμού Κομφιντούστρια στην Ιταλία. Έχετε το λόγο για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ πολύ και που οργανώσατε αυτή την τόσο σημαντική συνάντηση για τον ε, τουρισμό. Ε, ξεκινώ λοιπόν από αυτό που ελέγχθη, ότι ο τουρισμός είναι ένας από τους τουρισμούς, ένας από τους κλάδους οικονομίας ε, που έχει μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης, κυρίως μέσα σε ε, πέντε χρόνια 140 εκατομμύρια νέοι τουρίστες προέκυψαν και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον κλάδο μας. Ο τουρισμός ε, ε, κατέχει περίπου το 52% και Νομίζω ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να δούμε πώς αυτά επηρεάζουν την απασχόληση. Ο κλάδος που εκπροσωπούμε έχει αντιμετωπίσει μια σειρά πολλών προκλήσεων. Μεταξύ αυτών είναι η ψηφιοποίηση της αλυσίδας αξίας, τουλάχιστον όσον αφορά την ε, διανομή των προϊόντων και την τοποθέτηση των προϊόντων στην αγορά. Κατόπιν υπάρχει και ο ανταγωνισμός, εμφανίζονται νέοι παίκτες και αυτό που ενδιαφέρει είναι η σχέση ανάμεσα στο κόστος ε, και το τελικό προϊόν. Και τέλος υπάρχει και η εποχικότητα. Η Ευρώπη αναμφίβολα επ' αυτού θα πρέπει να μας βοηθήσει γιατί σε γενικές γραμμές η Ευρώπη είναι η περιοχή εκείνη όπου το εποχικό στοιχείο είναι ιδιαίτερα έντονο. Και ε, αυτό που ε, ευχόμαστε είναι να υπάρξει μια αλλαγή, αλλαγή της τάσης και των ε, καταναλωτών. Δηλαδή από ένα μοντέλο οικονομίας παροχής υπηρεσιών να πάμε όλο και περισσότερο σε μια οικονομία η οποία θα βασίζεται στο, στα βιώματα, να είναι ένας κλάδος με ιδιαίτερο επαγγελματισμό. Αυτό που εμείς θεωρούμε πολύ σημαντικό είναι να υπάρξουν επενδύσεις, να βελτιωθούν οι δυνατότητες που διαφαίνονται και αυτό σε τέσσερις κυρίως τομείς. Να στηριχθεί η επιχειρηματικότητα, η ψηφιοποίηση, η αηφορία και η καινοτομία. Αυτά είναι καθοριστικά στοιχεία για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα του τομέα. Εμείς ως ε, ε, οργάνωση θέλουμε να επιτύχουμε αυτή την ανάπτυξη όχι μόνο στον όγκο, αλλά κυρίως ε, στην ποιότητα, ποιοτική βελτίωση και αναβάθμιση. Για να προσελκύσουμε περισσότερες επενδύσεις, κρίνουμε ότι είναι καθοριστική σημασία να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τις, τα κονδύλια τα οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη διαθέτει στα κράτη-μέλη, να ε, γίνει κάποια έρευνα που ακριβώς πρέπει να γίνουν οι επενδύσεις, έτσι ώστε να γίνεται και καλύτερη χρήση των κονδυλίων. Παραδείγματο χάρη, υπάρχουν κονδύλια ε, που δίδονται για την ανάπτυξη των περιοχών και σχετίζονται με την πολιτιστική ανανέωση. Στην Ιταλία 32 δις 700 εκατομμύρια θα δοθούν ακριβώς ε, για την ε, βελτίωση και την προβολή του, ε, της τέχνης και του πολιτισμού. Η Επιτροπή έχει προτείνει να ενισχυθεί ο τομέας των μεταφορών με 400 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 17-20. Εμείς προτείνουμε από αυτό το ποσό 50 εκατομμύρια να δοθούν για την διασύνδεση των μέσων μεταφοράς. Ε, να σας πω το εξή ότι στην Ιταλία έχουμε 66 εκατομμύρια ταξίδια που έχουν σχέση με τουρισμό. Ένα άλλο θέμα αφορά στην ψηφιοποίηση. Στην Ιταλία έχουμε ένα πολύ μεγάλο χάσμα, έλλειψη ανταγωνιστικότητα στον τομέα αυτό και τα βασικά εμπόδια τα αναφέραμε. Ε, οι επιχειρήσεις έχουν, οι μικρομεσαίες κυρίες έχουν πολλά εμπόδια γιατί δεν έχουν και τα απαραίτητα κονδύλια για να εκπαιδεύσουν και το προσωπικό τους. Ως εκ τούτου πρέπει να τους διευκολύνουμε να έχουν καλύτερη πρόσβαση στην ψηφιοποίηση γιατί με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουν να έχουν και καλύτερη επαφή και με τους πελάτες αυτό που είναι σημαντικό είναι να δημιουργούνται οικονομίες ε, κλίμακος, ε, εποφελείς και κερδοφόρες ε, εταιρικέ σχέσεις. Υπάρχουν επαγγέλματα που αναδύονται σε μεγάλο βαθμό, είναι τα επαγγέλματα εκείνα τα οποία έχουν σχέση με την ψηφιοποίηση. Ω εκ τούτου θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε αυτέ τι ε, νέε ανάγκε. Εμεί κάναμε μια έρευνα στι επιχειρήσει ε, και πάρα πολλέ, παραδείγματο χάρη, ε, ασχολούνται με το web contest, με την επαγγελματική προβολή του. Εμεί, ως Ένωση έχουμε ένα εργαστήριο το οποίο βοηθάει και ασχολείται και με την αειοφορία που είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Ήδη σήμερα υπάρχουν 3 εκατομμύρια θέσει εργασία που σχετίζονται με την αηφορία και την βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά μισό λεπτό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι και η προστασία των δεδομένων, τα big data κυρίως. 9.000 ε, θέσει εργασία θα προκύψουν στην Ιταλία για την προστασία των δεδομένων, για την εκπαίδευση. Και κλείνω με αυτό. Εμείς είμαστε πεπισμένη ότι αυτή θα πρέπει να αφορά κυρίως τους νέους από 16 μέχρι 35 ετών. Σήμερα η οργάνωσή μας, η Φέντερ Turismo, είναι επικεφαλής σε δύο προγράμματα και Ευχαριστούμε τις Επιτρόπους Κώστα και Τίσεν γιατί εμείς ασχολούμεθα με δύο βασικά προγράμματα. Το ένα έχει σχέση με τη σταδιοδρομία και το επόμενο, το άλλο έχει σχέση με την επόμενη ε, γενιά τουρισμού. Στο δεύτερο κυρίως ο στόχος είναι να υπάρξει μια στρατηγική σχέση ανάμεσα στις επιχειρήσεις έτσι ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τουρισμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, Χίλια, ευχαριστούμε. Περνάμε στον επόμενο μας καλεσμένο, τον κύριο Τόμας Ράινχαρτ, που είναι, είναι διευθυντής ε, ε, των αερογραμμών της Ευρώπης και μάλιστα σίγουρα η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού έχει μεγάλο ενδιαφέρον για το τι συμβαίνει στον κλάδο σας και με ιδιαίτερη χαρά σας δίνω το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την παρουσία μας εδώ, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, εξοχότητες, κυρίες και κύριοι. Όντως, έχουμε καλή συνδεσιμότητα, θα έλεγα, με την Επιτροπή Μεταφορών, γιατί η συνδεσιμότητα είναι η λέξη κλειδί και πολύ μόδας για την Ευρωπαϊκή Αεροπορία και για πολλά άλλα θέματα και κλάδους. Και το θέμα της ε, συνδεσιμότητας είναι πολύ σημαντικό και στον τουρισμό. Οπότε θα έμεινω κι εγώ σε αυτό. Παίζει τεράστιο ρόλο η διασυνδεσιμότητα γιατί συνδέει τους ε, τουρίστες στην Ευρώπη. Σίγουρα ε, η, τα αεροπορικά εισιτήρια δεν ήταν ποτέ τόσο φτηνά όσο σήμερα και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από δύο μήνε όρτασε τα 25 χρόνια τη απελευθέρωση τη Ευρωπαϊκή Πολιτική Αεροπορία και μάλιστα το 1992 μια τετραμερή οικογένεια πηγαίνοντα από το Μιλάνο στο Παρίσι θα έπρεπε να πληρώσει 1.600 ευρώ και σήμερα η ίδια τετραμερή οικογένεια στην ίδια ε, πτήση θα πλήρωνε περίπου 100 ευρώ. Βλέπετε έχουμε τεράστια μείωση των τιμών χάρη στην απελευθέρωση ε, των υπηρεσιών στην πολιτική αεροπορία. Και οι αεροπορικές γραμμές προσπαθούν να κρατήσουν χαμηλά το κόστος για να μπορούν όλοι οι πολίτες να αγοράζουν σε, σε προσιτές τιμές αεροπορικά εισιτήρια. Και για να το εξασφαλίσουμε αυτό, θα επικεντρωθούμε σε τρία πράγματα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα, αλλά τα τρία είναι βασικά. Να δούμε πώς θα μειώσουμε τα τέλη αεροδρομίων που επιβαρύνουν τα αεροπορικά εισιτήρια και τις αεροπορικές εταιρείε και τους πελάτες ε, γι' αυτό θα πρέπει να μειώσουμε τα τέλη αεροδρομίου. Επίσης, να βρούμε καλύτερους τρόπους ε, ε, για ένα, ένα αέριο ευρωπαϊκό χώρο που θα είναι αποδοτικός ε, σε ό,τι αφορά το κόστος, οφέλους το κόστος και το όφελος και επίσης να περιορίσουμε τις απεργίες των ελεκτών ενέργειας κυκλοφορίας για να περιορίσουμε και τις ακυρώσεις πτήσεων. Επίσης, για τα τέλη της αεροπορίας, Σίγουρα το, η τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου σας αυξάνεται παρόλο που δεν το ξέρετε σε πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω των ε, ε, τελών ή των φόρων της αεροπορίας. Μερικές χώρες τις αποκαλούν περιβαλλοντικούς φόρους. Πάντως επηρεάζει άμεσα αυτή τη τιμή εισιτηρίου. Τώρα, για τα τέλη αεροδρομίου, πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε και μάλιστα την οδηγία για τα τέλη αεροδρομίου Ελπίζω να κάνει ό,τι μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να τηρήσει τις υποσχέσεις της και να αναθεωρήσει την οδηγία. Βέβαια δεν είναι σαφές ακόμη ε, πότε και αν η νομοθετική πρόταση θα εμφανιστεί εμπρόθεσμα, γιατί είναι λίγο αργά για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νέε νομοθετικέ προτάσει. Πάντω, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι τα τέλη αεροδρομίου ε, επιβαρύνουν κατά 20% τι αεροπορικέ εταιρείε ε, είναι το 20% του κόστους διαχείρισής τους ε, και επιβαρύνουν φυσικά αντίστοιχα το, την τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου. Και μάλιστα πριν από 20 χρόνια η τιμή του εισιτηρίου έχει μειωθεί κατά 20% ενώ οι τιμές, ε, οι, τα ποσοστά των τελών αεροδρομίου έχουν αυξηθεί κατά 80%. Επίσης, οι απεργίες των ελεκτών εναέρειας κυκλοφορίας. Πέρυσι ε, έγιναν πολλές τέτοιες απεργίες, ένα πολύ ακαθόδες ζήτημα και την τελευταία επταετία οι απεργίες αυτές των ελεκτών εναέρειας κυκλοφορίας προκάλεσαν τεράστιες ζημίες, έγινε κακή διαχείριση και κόστησαν περίπου 12 δισεκατομμύρια ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία και περίπου 140.000 θέσεις απασχόλησης. Όντως υπάρχει κόστος για τις εναέριες, ε, ε, για τις αεροπορικές εταιρείες λόγω των απεργιών και περίπου 60% του κόστους των 12 δισεκατομμύριων αυτών των απεργιών έπληξε τον τουριστικό κλάδο γιατί ο κόσμος θέλει να πάει διακοπές από το βορρά στο νότο ε, τα σχέδιά τους ακυρώθηκαν λόγω των απεργιών. Οπότε ακύρωνα, ακυρώνονταν οι πτήσεις, ακυρώνονταν τα ξενοδοχεία, δεν πήγαιναν στα εστιατόρια και έτσι επιδεινώθηκε η ανεργία στον τουριστικό κλάδο, κυρίως στις χώρες του Νότου, που ήταν οι χώρες προορισμού. Επίσης, οι απεργίες επηρεάζουν και την συνδεσιμότητα των τουριστών, ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη. Επίσης, τέλη αεροπορικής κυκλοφορίας. 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν η συνεισφορά των αεροπορικών εταιριών μόνο λόγω αυτών των ε, τελών ή φόρων αεροπορίας. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνονται οι πολίτε, πάντω το κόστο για τι αεροπορικέ εταιρείε είναι πολύ υψηλό. Και χώρε όπω η Σουηδία αποφάσισαν να θεσπίσουν ένα τέτοιο φόρο αεροπορία και τώρα έχουν συνειδητοποιήσει ποιο θα είναι ο αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο στην τοπική οικονομία. Θα το αρχίσουν να το εφαρμόζουν από τον Ιανουάριο. Η Ιρλανδία και η Ολλανδία κατήργησαν του αντίστοιχου φόρου ε, αεροπορία γιατί είδαν πόσο αρνητικέ είναι οι επιπτώσει του. Μέσα σε ένα χρόνο λοιπόν κατήργησαν αυτά τα τέλη και άνθισε ως εκ τούτου ο τουρισμός τους και αυξήθηκαν οι πτήσεις. Οπότε, όταν μιλούμε για τη διασυνδεσιμότητα, θα πρέπει να προσέξουμε αυτούς τους τρεις τομείς που σας ανέφερα. Και από την άποψη της διασυνδεσιμότητας ε, και των αεροπορικών μεταφορών, πιστεύω ότι μπορούμε να συνεργαστούμε και με, αντιμετωπίζοντας τα τρία αυτά προβλήματα, να βελτιώσουμε την διασυνδεσιμότητα στον τουρισμό. Σας ευχαριστούμε. Όπως είπατε, θα πρέπει να συνεργαστούμε. Γι' αυτό ακριβώς σας προσκαλέσαμε. Επόμενος ο μιλητής είναι ο κ. Πάτρικ Τόρεντ, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Περιφερειών για ανταγωνιστικό και βιώσιμο τουρισμό. Το τελευταίο διήμερο, μάλιστα, συναντηθήκαμε μαζί του, με τον κύριο Πάτρικ Τόρεντ τρει-τέσσερι φορές, οπότε ήδη είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις. Όχι μόνοι μας βέβαια, αλλά τώρα θα τις παρουσιάσουμε και μπροστά στους άλλους 300-400 συναδέλφους. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ που μας δίνετε το λόγο. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειών για έναν τουρισμό ανταγωνιστικό και βιώσιμο ε, το, είναι ένα δίκτυο το οποίο εκπροσωπώ και είναι μεγάλη τιμή που έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τους κοινούς μας στόχους. Στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε μια ευρωπαϊκή στρατηγική που θα έχει αηφόρο ανταγωνιστικότητα στο τουρισμό για ε, δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Ταγιάννη, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και όλες τις πολιτικές ομάδες, γιατί μας άνοιξαν την πόρτα, μας κάλεσαν εδώ, μας ε, κάλεσαν να συμμετάσχουμε για πρώτη φορά σε αυτή τη συζήτηση. Και αυτό για μας είναι ιστορική στιγμή, διότι σήμερα πλέον στο μέσο της ανάπτυξης στην Ευρώπη, σε αυτή την προβληματική θεματική μπαίνει στην κεντρική θέση το, ο τουρισμός και όλοι χαιρόμαστε γι' αυτό. Το 2017 κλείνουμε 10 χρόνια ως Ευρωπαϊκό Δίκτυο που εκπροσωπούμε τις ε, περιοχές που είναι μέσα στους 20 πρώτους τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη και γιορτάζουμε λοιπόν αυτή τη μοναδική ευκαιρία ε, για τον αηφόρο τουρισμό για την ανάπτυξη. Έχουμε την ευκαιρία να συμβάλλουμε στους στόχους του αηφόρου ανάπτυξης χάρη ε, σε αυτή την θεματική χρονιά που κήρυξαν τα Ηνωμένα Έθνη. Η Ευρώπη είναι ο πρώτος τουριστικός προορισμός παγκοσμίω. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την ηγετική θέση, να καταβάλουμε μεγαλύτερη προσπάθεια και περισσότερες επενδύσεις. Καλύτερες επενδύσεις, ποιοτικότερο προϊόν, ποιοτικότερο προϊόν και να αξιοποιήσουμε το 2018 για τη δημιουργία ποιοτικού πολιτιστικού προϊόντος, να επενδύσουμε στην καινοτομία, στην έρευνα, στο να δώσουμε τις δυνατότητες στους επαγγελματίες του κλάδου να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους, να επενδύσουμε στις ευφυείς αγορές. Δεν μπορούμε να ε, ε, διαχειριστούμε αυτό που δεν μπορούμε να μετρήσουμε, άρα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στις μετρήσεις. Το 2018 θα είναι και το έτος τουρισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας και γι' αυτό προτείνουμε να υπάρξει εταιρικός, κοινωνικός διάλογος, ευρωπαϊκός διάλογος για ε, ε, να συμβαδίσουμε. Ε, περισσότερος διάλογος για την προώθηση του πολιτισμού και για να καταστούν οι τουριστικοί προορισμοί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κίνα αηφόροι, βιώσιμοι. Από τον Απρίλιο στη Βαρκελόνη ε, θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις, μια πολύ σημαντική συζήτηση για την κοινωνική πολιτιστική εργασιακή χρησιμότητα του τουρισμού. Και όλες αυτές οι συζητήσεις θα τροφοδοτήσουν το γενικότερο διάλογο. Μιλούμε για τις 19 Απριλίου στη Βαρκελόνη και είστε όλοι προσκεκλημένοι. Το δίκτυό μας επίσης προτείνει περισσότερες επενδύσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και καινοτόμων τουριστικών εμπεριών οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων να παρακολουθήσουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών, να ερευνήσουν τα big data για να καταλάβουν τι επιθυμούν οι καταναλωτές και να ε, τους προσανατολίσουν καλύτερα στην αντίστοιχη ε, προσφορά, να διαμορφωθεί η ζήτηση περισσότερη και καλύτερη, να αξιοποιηθούν όλα τα μέσα τα τεχνολογικά ε, για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε και με τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις startups, τις επιχειρήσεις τεχνολογίας για να διαμορφώσουμε καλύτερο προϊόν, ποιοτικότερο προϊόν. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για την ψηφιοποίηση στο πλαίσιο της έξυπνης ε, καινοτομία για τον, ε, για τον κλάδο αυτό. Οκτώ περιφέρειες θα προωθηθούν για να επενδύσουν ερευνητικά προϊόντα, ερευνητικές δραστηριότητες τεχνολογικών προϊόντων. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε το ΕΦΣΥ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, για να έχουμε μια στέρεα επενδυτική πλατφόρμα ε, μέσα στην, από την οποία θα βρίσκουν χρηματοδότηση οι περιφέρειες για, θέματα, για τουριστικά σχέδια. Δεν είναι εύκολο, μπορούμε μαζί να νικήσουμε και ε, καλούμε όλους να συμμετάσχουν σε αυτό το εργαλείο ε, χρηματοοικονομικής μηχανικής. Μπορούμε να εμπλουτίσουμε αυτή τη συζήτηση ε, για τα ευρωπαϊκά κονδύλια μετά το 2020. Να υπάρξει μια γραμμή στον προϋπολογισμό πιο ορατή και καλύτερα προσβάσιμη για τον τουρισμό. Είμαστε στη διάθεσή σας για να αναπτύξουμε μαζί μια νέα στρατηγική τουρισμού στην Ευρώπη προ όφελο των ε, επικρατιών, των περιφερειών, των περιοχών, των επιχειρηματιών, των πολιτών, ε, των κοινωνιών αλλά και των φιλοξενούμενών μα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα ξεκινήσαμε Ξεκίνησε και η Επιτροπή των Περιφερειών τις συνεδριάσεις της και της εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου. Ε, πρέπει η συνεργασία να είναι περισσότεροι και περισσότερο μπορούν να οργανωθούν σε διάφορα επίπεδα και εδώ στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο και αλλού ενίοτε θα ήταν πολύ χρήσιμο να μιλήσουμε και για το τουρισμό στη Σύνοδο της Ολομέλειας στο Στρασβούργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να καλωσορίσω θερμά την κυρία Λούρια Κεβάρα Μάντσο, τη νέα πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του WTC, του Παγκοσμίου Συμβουλίου Τουρισμού. Οι μεγαλύτερες οργανώσεις στον τομέα του τουρισμού είναι η Παγκόσμια Οργάνωση Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών και το WTTC, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού. Και η, η κυρία Γκεβάρα Μάντσο είναι πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος. Ήσασταν στο Μεξικό και τώρα είστε εδώ στην Ευρώπη, στην καρδιά των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων για να πάρετε το λόγο εκ μέρου του Παγκόσμιου Συμβουλίου Ταξιδιών και Τουρισμού. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους σας. Ε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ταγιάννη. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό το ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ και ε, όταν ανακοινώθηκε ότι θα οργανωθεί αυτή η συνάντηση. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ. Όπως είπε και ο πρόεδρος μας, τώρα έχω το άλλο ρόλο το, του, της Διευθυνούσης ε, Συμβούλου του Παγκόσμιου Οργανισμού ε, Τουρισμού. Όπως αναφέρθηκε λοιπόν, ο τουρισμός και τα ταξίδια ε, καλύπτουν περίπου το 10% του ΑΕΠ. Είναι η μία από τις δέκα θέσεις, κάθε δέκατη θέση στις στην την απασχόληση θα προκύψουν και πάρα πολλές άλλες θέσεις απασχόλησης. Εμείς ε, προσφέρουμε περίπου ένα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Είναι το 10% του ΑΕΠ στην Ευρώπη. Και αυτό σημαίνει 36 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης που εξαρτώνται από τα ταξίδια και τον τουρισμό. 72 δις επενδύσεων. Αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός. Τα ταξίδια και ο τουρισμός συμβάλλουν περισσότερο στο ΑΕΠ στην Ευρώπη από άλλους τομείς. Και θα ήθελα να σας αναφέρω ορισμένα παραδείγματα. Εμείς απασχολούμε τρεις φορές περισσότερους από ότι ε, οι τράπεζες στη Γερμανία απασχολούμε επίσης ε, ένα μεγάλο αριθμό ατόμων στη Γαλλία, ε, περίπου τετραπλάσιος ο αριθμός των δικών μας απασχολούμενων από ότι στις τράπεζες τα επόμενα χρόνια θα δημιουργηθούν πάνω από 5 εκατομμύρια θέσεις απασχόληση στην Ευρώπη. Όμως ε, χρειάζονται πολλά πράγματα. Και ένα από αυτά έχει συζητηθεί. Χρειαζόμαστε επενδύσεις. Προβλέπουμε 2,13 ευρώ θα επενδυθούν στην Ευρώπη τα επόμενα 10 χρόνια. Ε, όμως ε, για ευφυείς επενδύσεις χρειαζόμαστε περισσότερη τεχνολογία και καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ε, πρέπει να σπάσουν οι φραγμοί για την βελτίωση των επενδύσεων ε, να υπάρχει και το σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο. Ο στόχος βέβαια είναι να υπάρχει ποιότητα στον τουρισμό στις θέσεις απασχόλησης και είναι και πολύ σημαντικό να βλέπει κανείς και τα ε, συστήματα καινοτομίας ε, για να μπορεί να στηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις ε, για τον τουρισμό. Οι άνθρωποι πρέπει να ταξιδεύουν. Αυτό αναφέρθηκε ήδη. Αλλά η Ευρώπη είναι και παγκόσμιο ηγέτη στη μετακίνηση ατόμων. Γνωρίζουμε ότι υπήρξε δυσκολία λόγω του προσφυγικού. Ο δικός μας οργανισμός ασχολείται, γνωρίζει πολύ καλά τις εξωτερικές πιέσεις. Αλλά παράλληλα πιέζουμε τους ε, Ευρωπαίους ηγέτες ε, να πλουστεύσουν τις διαδικασίες για τις θεωρήσεις, κυρίως για αυτούς που θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη για σύντομες παραμονές. Και θέλω να πω ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να βρουν ε, μια ρεαλιστική λύση που θα ωφελεί τους περισσότερους Ευρωπαίους πολίτες. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει το θέμα της, ε, των θεωρήσεων, ε, κυρίως σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Χρειαζόμαστε λοιπόν φόρο ανάπτυξη. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται η αξία που προσφέρουμε και ο τοπικός σχεδιασμός ε, εξισορροπεί τις ανάγκες και της τοπικής κοινωνίας και του τουρισμού. Επ' αυτού πρέπει να συνεργαζόμαστε. Το Δεκέμβρη του 2013 θα είμαι στη Βαρκελόνη και εκεί θα αναζητήσουμε κάποιες μελέτες που αφορούν στο overcrowding και το πώς μπορούμε να χειριστούμε καλύτερα ορισμένους προορισμούς. Πρέπει να προστατεύουμε καλύτερα τους πόρους μας αλλά επίση και το όφελο που προκύπτει για τους πολίτες μας. Εάν τα καταφέρουμε όλα αυτά, τα ταξίδια και ο τουρισμός θα φτάσουν σε πάνω από 5 εκατομμύρια θέσει απασχόληση, ε, και ε, αντίστοιχα θα αυξηθεί και το ποσοστό στο ΑΕΠ. Είναι σημαντικό οι θέσει απασχόλησης να υπάρξουν σε όλους τους ε, τομείς, να αφορούν κυρίως τους νέους και τις γυναίκες και να υπάρχουν θέσεις σε όλες τις περιοχές. Κυρίες και κύριοι, είναι σαφές ότι τα ταξίδια και ο τουρισμός είναι η καλύτερη δυνατότητα για να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση. Όσον αφορά στον ιδιωτικό τομέα, θέλω να σα πω ότι εμεί είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σα. Μπορούμε να καθορίσουμε από κοινού τα θέματα που απασχολούν εμά και του πολίτε μα. Σα ευχαριστώ πολύ για την ε, υποστήριξή σα και χαίρομαι που οργανώσαμε αυτή την ε, εκδήλωση. Σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, φτάσαμε εσείς στις 5.30. Έχετε όλη την ημερήσια διάταξη της διάσκεψης υψηλού επίπεδου και ξέρετε το πρόγραμμά της. Πρέπει να περάσουμε αμελητή στη συνέχεια, στα, σε επόμενες δύο στρογγυλές τράπεζες. Η μία θα διεξαχθεί στην αίθουσα αυτή και η δεύτερη στρογγυλή τράπεζα στη διπλανή αίθουσα την 3C50. Ακολουθήστε την κυρία με την αφίσα που δείχνει τον αριθμό της αίθουσα. Ακολουθήστε την. Εκεί θα γίνει το δεύτερο πάνελ. Και τα δύο πάνελ είναι πολύ ενδιαφέροντα. Με, θα γίνουν με καλεσμένους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπουργού από τα κράτη-μέλη και φυσικά και ευρωβουλευτές. Η κυρία Κλάουντια Μοντέρο Ντιαγκιάρ, ευρωβουλευτής, θα είναι μία από τις ομιλήτριες στον επόμενο γύρο, στο, στην επόμενη στρογγυλή τράπεζα, οπότε κυρία Ντιαγκιάρ παραμείνετε στην αίθουσα. Όσοι θα παρακολουθήσουν την άλλη στρογγυλή τράπεζα, ας μεταβούν στη διπλανή αίθουσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ που συντώνησα αυτό το τμήμα της συζήτησης.